εκείνες οι περιοχές που μπορεί να χάσουν το καθεστώς τους, θα, για αυτές τις περιοχές θα προβλεφθεί ε, μία ειδική περίοδος μετάβασης. Ευχαριστώ, Επίτροπε, λέει Πρόεδρος. Τελειώνει η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε για το σημείο αυτό σε δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, στην ε, Μίνη Ολομέλεια. Έχουμε ακόμα ένα σημείο στη μερίσια διάταξη την έκθεση Richard Ashworth «Απλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής». Έχει το λόγο εισηγητής. Ε, Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, Βρισκόμαστε στα πρώιμα στάδια της συζήτησης που θα οδηγήσουν στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2012. Σε αυτή την έκθεση πρότεινα ορισμένες αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ. Καθίσταται σαφές ότι η γεωργική ομιχανία θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει για να αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις των καιρών μας, αλλά και τους μεταγενέστερους καιρούς δηλαδή η διατροφική ασφάλεια, η ε, μεταβλητότητα της αγοράς, οι κλιματικές αλλαγές και οι ανάγκες να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες έτσι ώστε να αποδώσουμε τα δημόσια αυτά αγαθά. Η ΚΑΠ θα πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές, αλλά καθίσταται σαφές ότι και ο τρόπος εφαρμογής της ΚΑΠ θα πρέπει να αλλάξει Ορίζοντας αυτές τις αρχές που διέπουν την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Αυτό θα γίνει αργότερα. Αυτό που πρότεινα όμως είναι δύο βασικά ζητήματα. Καταρχήν η ΚΑΠ να είναι απλούστερη, δικαιότερη και πιο διαφανής και δεύτερον ότι το πολιτιστικό υπόβαθρο της ΚΑΠ θα πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε η μελλοντική μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ να λαμβάνει υπόψη τις εκβάσεις και να μην είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική. Τέσσερις είναι οι τρόποι για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Να διασφαλίσουμε ότι οι απαιτήσει είναι αναλογικές με τον αποτιμόμενο κίνδυνο. Δεύτερον, να εναρμονίσουμε τα κριτήρια εποπτείας και να μην υπάρχει επικάλυψη ε, εποπτείων. επίσης να έχουμε μεγαλύτερη ε, εμβέλεια για την αυτοπιστοποίηση και τέταρτον οι κυρώσεις κατά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να είναι αναλογικές με το βαθμό της ε, παράβασης και να μην ε, είναι καταποκοπήν κυρώσεις όπως ισχύουν στην περίπτωση που οι παραβάσεις, για τις παραβάσεις δεν είναι υπέτη η γεωργή. Ένας στόχος της ΚΑΠ θα έπρεπε να είναι να βοηθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τη βιομηχανία να ε, προσαρμοστεί στις νέες αυτές αλλαγές. Γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή του πολιτιστικού μας υποβάθρου. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο ε, ευέλικτη προσέγγιση. Επίσης, να γίνονται περισσότερες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους βιομηχανικούς φορείς και να έχουμε καλύτερη αποτίμηση των επιπτώσεων του, των προτινόμενων κανονισμών οι οποίοι θα πρέπει να είναι πιο εύκολα ερμηνευόμενοι. Επίσης, θα πρέπει να δείξουμε ότι πραγματικά παραδίδουμε δημόσια αγαθά, μειώνοντας το κόστος της βιομηχανίας για συμμόρφωση και έτσι ώστε να διαχειριστούμε αποδοτικά τη βιομηχανία αυτή. Η έκθεση ορίζει αρκετούς τρόπους για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ashworth. Έχουμε αρκετούς ομιλητές που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο. Η κυρία Εσάια είναι η πρώτη. Ευχαριστώ. Σε σχέση με το διοικητικό φόρτο θα πρέπει να μειωθεί για τους γεωργικούς παραγωγούς ε, κατά τους τρόπους που ανέφερε ο εισηγητής. Ευπρόσδεκτα τα μέτρα που προτείνει πολλοί γεωργοί θεωρούν στην ουσία ότι είναι εγκληματίες και έτσι τους αντιμετωπίζουμε με αυτό το γραφειοκρατικό φόρτο. Η ΚΑΠ θα πρέπει να είναι πιο απλουστευμένη και παράλληλα όταν η αγορά αλλάζει και όταν ε, υπάρχει λιγότερος προστατευτισμός ως προς τις αγωγές θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και συγκεκριμένους μηχανισμούς όπως το μηχανισμό παρέμβασης ή τις επιδοτήσεις κατά τις εξαγωγές. Αυτά θα πρέπει να αναθεωρηθούν κατά το μέλλον, το οποίο δεν είναι καθόλου απλό, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό που να προσωμιάζει με τις ποσοστώσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Τσαμπάντη. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί οι προτάσεις και η φιλοσοφία της έκθεσης είναι αξιέπαινες. Έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τους ε, πραγματικά ενεργούς γεωργούς, αυτούς που καλλιεργούν τη γη. Ακριβώς γι' αυτό αξίζει συγχαρητήριον η πρόταση. Στο μέλλον η ΚΑΠ θα πρέπει να ξεφορτωθεί τις ε, τομεακές διαφορές και θέλω να τονίσω ότι υπάρχει διάκριση εναντίον των νέων κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό να απλουστευτούν οι κοινοτικοί κανόνες και να εφαρμοστούν σωστά στα κράτη-μέλη. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πριν δύο χρόνια το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα κανονισμό και κατέστη υποχρεωτικό το να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή των ζώων. Σε κάποια κρατημέλη που δεν υπήρχαν ε, επιδοτήσεις, οι κτηνοτρόφοι δεν ήξεραν τι να κάνουν οι υπερβολικοί, οι κανόνες και η γραφειοκρατία μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η έκθεση είναι πολύ, τόσο σημαντική. Ο κύριος Ντόρφμαν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Άσχορτ, για αυτήν την εισήγηση πιστεύω ότι η ΚΑΠ είναι μια πολιτική η οποία λειτουργεί. Καμιά φορά όμως υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και για αυτό αφορά διάφορες ε, πλευρές της κοινή ε, αγροτικής πολιτικής. Ας μην ξεχνούμε τις μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τεράστια γραφειοκρατία υπάρχει και για, σε ό,τι τις αφορά πρέπει να βρούμε μια καινούρια μέθοδο λοιπόν για να μπορέσουμε με αυτήν τη νέα μέθοδο η οποία θα επιτρέψει μια απλούστευση για τις επιχειρήσεις οι οποίες κινούνται με μερικές χιλιάδες ευρώ μόνο να μπορούν να δράσουν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τον γενικό μας στόχο που είναι ότι δεν θα πρέπει να ε, υπάρχουν απάτες. Ευχαριστώ. Η απλούστευση της ΚΑΠ, ε, όπως προτείνεται από αυτή την πρόταση, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και το μοναδικό αυτής της έκθεσης είναι ότι εξετάζει τα πάντα από τη σκοπιά των γεωργών. Επίσης, το, τα χρήματα προς τους γεωργούς είναι το μέσο. Ο στόχος είναι να υλοποιηθούν οι πολιτικές. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μέσων και στόχων. Πρέπει να αλλάξουμε εντελώ τις συμπεριφορές. Οι πελάτες που είναι γεωργοί σε σχέση με τις agencies, με τις υπηρεσίες, δεν θα πρέπει να πέφτουν θύματα της γραφειοκρατίας. Η Κομισιόν θα πρέπει να εκπονήσει ένα κανονισμό που θα προβλέπει ότι και οι agencies θα πληρώνουν πρόστιμα εάν δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και θα πρέπει να πηγαίνουν και στα δικαστήρια. Στην Ουγγαρία δεν υπάρχει πια περίπτωση αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει σημασία είναι η απλούστευση της ΚΑΠ. Είναι πολύ καλή ιδέα. Κανένας θα μπορούσε να αντιταχθεί στη μείωση του διοικητικού κόστους των οργάνων εποπτείας και το, του χρόνου εργασίας των αγροτών. Αυτή είναι εξαιρετική ιδέα θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι εφαρμογής. Καταρχήν υπάρχουν τομείς παραγωγής ε, για τις οποίες είναι δύσκολο να υπάρχουν επιδοτικοί μηχανισμοί, παραδείγματος χάρη στον τομέα των καπνών. Ως προς την διατήρηση της παραγωγής στις περιφέρειες όπου υπάρχουν δυσκολίες, δυσχέρειες γενικότερα, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί επιδότησης της παραγωγής, αλλά εξειδικευμένοι μηχανισμοί. Όπως είπε ένας από τους προλαλήσαντες, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η ΚΑΠ στο μέλλον θα πρέπει να είναι μία απλουστευμένη ε, πολιτική, διαφανής και αποδοτική. Για να φτάσουμε στην απότερη απλούστευση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ΚΑΠ θα πρέπει να είναι πιο απλή, πιο διαφανής και πιο κατανοητή στο μέλλον. Αυτό είναι το μήνυμα της έκθεσης του κυρίου Ashworth και είναι πολύ σωστό. Η έκθεσή μας θα πρέπει να ενθαρρύνει την Κομισιόν να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω απλούστευση της ΚΑΠ. Αυτό είναι προς το συμφέρον των γεωργών μας, οι οποίοι θα κέρδιζαν χρόνο καταρχήν. Νομίζω ότι κερδίζοντας τέτοιο αυτό το χρόνο θα τους έδινε περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με την βασική τους δραστηριότητα, που είναι η καλλιέργεια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είναι αυτό η προτεραιότητα της Κομισιόν. Δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Ξαναδίνω το λόγο στον Επίτροπο που θα κλείσει και τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, η απλούστευση και η σωστή διαχείριση είναι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Άσχοτ για την εξαιρετική εισήγηση του σε έναν τομέα ο οποίος ε, αντιμετωπίζεται με θάρρος και πρόκληση. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους γεωργούς. Ε, το, πολλές φορές έχουν ε, οι γεωργοί το λόγο για την κύρια αγροτική τους διαδικασία. Υπάρχει ένας τομέας μεγάλης ανησυχίας λοιπόν για τους γεωργούς ο οποίος απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτή την έκθεση υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις και πολλές προτάσεις οι οποίες επιτρέπουν στην Επιτροπή να ανανεώσει την κοινή αγροτική πολιτική θα ήθελα να υπογραμμίσω το σημείο όπου γίνεται σύσταση στην Επιτροπή για το ε, φόρτο της γραφειοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο παρεμποδίζει τις ε, δραστηριότητες των ε, γεωργών και η απλούστευση είναι κάτι το οποίο το έχει αναλάβει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια διαδικασία την οποία ήδη ακολουθούμε και πέρα από αυτό υπάρχει μια γενική περισσότερη συλλογή για την ε, όλη διαδικασία που θα διέπει την κοινή αγροτική πολιτική στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί από κοινού για να έχουμε μια αποτελεσματικότητα στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη μείωση του φόρτου ενώ θα υπάρχει μια υψηλή προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής, γιατί η γεωργία είναι ένας δοτικός τομέας. Ε, πρέπει επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία, ήθελα να το αναφέρω αυτό και προηγουμένως, ότι σε σχέση με την απλούστευση. Δεν θα πρέπει η απλούστευση να γίνεται σε βάρος των προκλήσεων που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματο χάρη η ιχνηλασιμότητα. Πέρσι είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ως προς αυτό το πρόβλημα. Ε, ε, υπήρξαν ορισμένες ε, επιδημίες οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταργήσουμε το πρόβλημα απλώς της συχνηλασιμότητας γιατί υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία στην οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εάν απλουστεύσουμε τις διαδικασίες πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσουμε όμως ορισμένους κανόνες μέχρι πέρατος. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να μας βοηθήσουν να είμαστε προσεκτικοί, να να μην καταργήσουμε και τα θετικά μαζί με τα αρνητικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πέρα στη συζήτηση οι ψηφοφορίες θα γίνουν σε δύο εβδομάδες από σήμερα στην Ολομέλεια των Βρυξελών. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο το πρωί στις 20 ε, Απριλίου Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 και από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις ε,